Εξηγήσεις ψήφου πριν τη διακοπή. Για τον διορθωτικό προϋπολογισμό, το λόγο έχει η κυρία Ντότς. Κύριε Πρόεδρε, εκτιμώ πολύ και εσάς ως πρόσωπο και τις ικανότητές σας. Όμως σήμερα διαμαρτύρομαι. Δώσατε σε πολλούς τον λόγο, όπως Φόξ, Γκόλνις και άλλους. Και εγώ ζήτησα τον λόγο για το χρονοδιάγραμμα των περίοδων συνόδου για σημαντικό θέμα. Παρακαλώ να εξετάσετε την τροπολογία 4, την οποία απορρίψαμε μένα, αλλά το θέμα είναι θέμα αρχής. Μήπως και αυτή είναι μη παραδεκτή, διότι στην συνθήκη δεν λέει 12 ε, περίοδοι συνόδου τον χρόνο, αλλά 12 μηνιαίες περίοδοι συνόδου τον χρόνο και η ε, τροπολογία Fox είχε τον στόχο να συγχωνεύσει την ε, περίοδο συνόδου του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου. Και παρακαλώ να διευκρινιστεί ότι κάτι τέτοιο είναι σαφώς παράνομο. Κύριε Πόσελτ, αυτό το θέμα το ψηφίσαμε ήδη. Δεν μπορούμε να ξανανοίξουμε το θέμα αυτό. Να είστε βέβαιος πάντως ότι όλες αυτές οι τροπολογίες επί το χρονοδιαγράμματος έτυχαν προσεκτικής εφαρμογής από τον Πρόεδρο. Προσεκτικής εξέτασης, συγγνώμη. Sí, señora σλίτερ, Señor σλίτερ. Κυρία Σλέιτερ. Ο κύριος, συγγνώμη. Σλέιτερ. Λειτουργεί καταρχήν το μικρόφωνο. Ο Επίτροπος μας ενημέρωσε αμέσως πριν την ψηφοφορία για ένα θέμα και ήθελα να ζητήσετε τα στατιστικά δεδομένα που λέει ότι διαθέτει για να δικαιολογήσει, να αιτιολογήσει μάλλον την ε, δήλωσή του ότι αυτό είναι υποφελές και ε, ωφέλιμο για τους καταναλωτές. Διότι τα πρόσθετα συστατικά για τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα σε λουκάνικα και άλλα προϊόντα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ωφελήσουν τους καταναλωτές με τη νέα χρήση που προτείνεται. Που, επίσης ο Επίτροπος έκανε τη σύγκριση με τον κοιμά. Ξέρουμε όμως ότι τα πρότυπα υγιεινής για τον κοιμά δεν είναι τα ίδια με τα επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος. Άρα και οι δύο δηλώσει του Επιτρόπου χρήζουν αιτιολόγηση. Ανθισβητώ εγώ την ορθότητά του. Πιστεύω λοιπόν ότι έχει διπραχθεί σοβαρό σφάλμα μέσω πριν την ψηφοφορία και θα ήθελα να συντάξετε επιστολή προ τον Επίτροπο ώστε να αιτιολογήσει ακριβώ τι δηλώσει του. Ευχαριστώ. Δεν φτάσαμε ακόμη στο σημείο αυτό, κύριε Σλίτερ. Είμαστε στι επεξηγήσει ψήφου. Επεξηγήσει ψήφου για το διορθωτικό προπολογισμό. Το λόγο έχει η κυρία Ντότ. Αποσιάζει la la η κυρία Ντότς. Το λόγο κύριο κύριος Φάσμπολ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ κατεψήφισα ε, την έκθεση. Δεν είμαι υπέρ της ιδέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα σε περίοδο κρίσεως να αυξάνει τις δαπάνες. Ούτε είμαι υπέρ των αυξήσεων των επιδομάτων για συνεργάτες περισσότερα δηλαδή από όσα έχουμε ήδη. Οι βουλευτές υποτίθεται θα έπαιρναν 1500 ευρώ παραπάνω ανά μήνα για τους συνεργάτες και αυτό σημαίνει πολλά εκατομμύρια εν τέλει ανά έτος. Και μας επικρίνει ολόκληρη κοινή γνώμη διότι διαθέτουμε τέτοιου είδους ποσά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει ολόκληρη Ευρώπη να κάνει οικονομήσεις και εμείς επομένως το ίδιο. Ευχαριστούμε κύριε Φάσμον. Ο κύριος Λιμπεράτσκι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σε αντίθεση με τον προλαλήσαντα ψήφισα υπέρ του διορθωτικού προϋπολογισμού γιατί δεν είναι μόνο λογιστική η διόρθωση, έχει βαθιά σημασία η διόρθωση αυτή. Και μάλιστα απορρέει από τις νέες μας αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε πια ε, ένα σώμα με νομοθετικές εξουσίες. Αυτό περιμένουν και από εμά οι ψηφοφόροι μας να καταφέρουμε να διορθώσουμε τους προϋπολογισμούς που μας υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουν οι πολίτες μας να είμαστε σε θέση να διορθώσουμε τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου και να υποστηρίξουμε τους ε, ε, επιτρόπους που υποστηρίζονται από πολυάριθμο προσωπικό. Εμείς έχουμε ελάχιστους βοηθούς. Δεν είναι θέμα οικονομίας, αλλά είναι απάντηση και ανάληψη των νέων μας καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή μας για την καταπληκτική του έκθεση και ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Λιμπεράτσκι. Περνάμε τώρα στην ε, έκθεση Μικολάσικ για τις μεταμοσχεύσεις. Πρώτος επεξήγηση ψήφου θα κάνει ο κύριος Μπιγκένιν. Σωστά. Σωστά Μπιγκένιν. ¿Y por qué no habla? No, no ha sentido. Κύριε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας πω ότι για την έκθεση περί μεταμοσχεύσεων και επειδή έχει να κάνει με την έλλειψη, την ανεπάρκεια οργάνων και τη χρήση τους, ε, ψήφισα διότι ελπίζω ακριβώς ότι η έκθεση για την ποιότητα των οργάνων θα επιτρέψει τα κράτη-μέλη να εναρμονίσουν τα κριτήριά τους Επίση ότι εδώ θα διαμορφώσουμε σύστημα που θα μα επιτρέψει να υποφεληθούμε και στο μέλλον στη χώρα μου. Τη Βουλγαρία υπάρχουν 35%, 35 μάλλον ε, αναλογικά λιγότεροι, 100 λιγότεροι δωρητέ από ό,τι στην Ισπανία λόγου χάρη. Πρέπει λοιπόν να ενημερωθούν ε, επαρκώ οι πολίτε για να βελτιωθεί όλη η διαδικασία μέχρι να φτάνουμε στη μεταμόσχευση. Αν δεν υπάρχουν δωρητέ, δεν έχουμε και αρκετέ μεταμοσχεύσεις. Επίσης χρειάζονται βάσεις δεδομένων, απαραίτητα στοιχεία. Στη Βουλγαρία μας λείπουν πολλά από αυτά για τις μεταμοσχεύσεις, καθώς και η αγωγή η μεταγχειρητική δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Ούτε υπάρχουν και μονάδε στα νοσοκομεία που να εξασφαλίζουν την παρακολούθηση των ασθενών. Ελπίζω λοιπόν ότι η έκθεση και ο θα μα παροτρύνουν να δράσουμε περισσότερο. Η κυρία Η κυρία έχει το λόγο ka mina hääletasin <clears throat> antud raporti poolt sest sellega Υπερψήφισα την έκθεση διότι καθιερώνει ομοιόμορφες απαιτήσει σε όλες τις χώρες μέλη σχετικά με τα ποιοτικά επίπεδα των οργάνων κάτι το οποίο θα αυξήσει την προστασία και των δωρητών οργάνων και των απολυπτών οργάνων και θα σημάνει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας των εγχειρήσεων που εν τέλει αφορούν 56.000 πρόσωπα το χρόνο. Κυρία Και εγώ χαίρομαι για ε, την πρόταση. Εάν μπορούμε να φροντίσουμε να είναι διαφανές το σύστημα και ξεκάθαρο των μεταμοχεύσεων, θα είναι σημαντική ωφέλεια για 56.000 ε, Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι αναμένουν ε, να ευρεθεί δωρητής γιατί βεβαίω η σπάνιση των οργάνων οδηγεί και σε άλλα προβλήματα όπω αύξηση τη εγκληματικότητα. Εγώ πιστεύω ότι η πρόταση αυτή μπορεί να δημιουργήσει ένα σύστημα ε, διασύνδεση με του δωρητέ που θα είναι και σημαντικό για την ασφάλεια των μεταμοχεύσεων. Ο Κάστλερ. Συγχαίρω τον κύριο Μικολάσικ για την εξαίρετη εργασία του. Εγώ υπερψήφισα Πρόκειται για σημαντική ημέρα σήμερα αφού ε, οι ομοιόμορφες αυτές απαιτήσεις, οι ενίες αυτές απαιτήσεις φροντίζουν, εξασφαλίζουν δηλαδή την ποιότητα των μεταμασχεύσεων. Και ελπίζω ότι θα οδηγήσουν και σε απλούστευση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών. Χαίρομαι λοιπόν που υπερψηφίστηκε η πρόταση αυτή με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ καλωσορίζω αυτή την έκθεση και τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την δωρεά οργάνων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα όργανο, υπάρχει, καλό είναι να χρησιμοποιηθεί για την ασφάλεια των ζώων των πολιτών. Και βεβαίω σε όλες τις χώρες χρειάζονται μέτρα τα οποία είναι λογικά και να μπορούν να υλοποιηθούν ευέλικτα. Εδώ να εκφράσω την προσωρική μου στήριξη για ένα σύστημα όπως αυτό που περιγράφεται στον κανονισμό και όχι ένα σύστημα Διότι το 80% των Ευρωπαίων πολιτών λένε ότι στηρίζουν την δωρεά των οργάνων, ενώ και για το 12% πρέπει να καλύψουμε το χάσμα. Ήδη 25 άνθρωποι στην δική μου εκλογική περιφέρεια, Πρόεδρε, ε, έχασαν τη ζωή του γιατί ακριβώ δεν μπορούσε να βρεθεί δωρητή για τη δική του μεταμόσχευση. Ήδη στην εκλογική μου περιφέρεια, στα νοσοκομεία υπάρχει πολλοί κόσμο που περιμένει και υπάρχουν ευρωπαϊκέ ανάγκε εδώ και για την ε, μεταναμόσχευση καρδιά. Εδώ λοιπόν να δώσουμε την ευκαιρία στου ασθενεί μα να λάβουν την ε, αγωγή και την περιθάψη που χρειάζεται. Είναι ένα θέμα ζωή. Ο κύριος, η κυρία Μαλόν Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή και είμαι ευγνώμων διότι υπερψηφίστηκε με τόσο μεγάλη πλειοψηφία. 56.000 Ευρωπαίοι σήμερα περιμένουν ένα κατάλληλο συμβατό όργανο για μεταμόσχευση, ούτως ώστε να μπορέσουν να ζήσουν και με κάποια ποιότητα ζωής. Ήταν κατεπήγον να κάνουμε ενιαία πρότυπα, να τα βελτιώσουμε και να βελτιώσουμε σε όλη την Ευρώπη την καλύτερη πρόσβαση στα όργανα. Ευχαριστώ. Ο Ζέμκε. Και εγώ υποστήριξα αυτό το έγγραφο. Νομίζω ότι πρόκειται για να βήμα σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα όμως να καταστήσω σαφές ότι είναι ένα πρώτο βήμα αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε περισσότερους δωρητές, αυτό που χρειάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σύστημα καλύτερης πρόληψης των ασθενειών και καλύτερης ενημέρωσης των ασθενών και των πολιτών μας γενικότερα. Γιατί αυτά είναι προαπαιτούμενο για να μην χρειαζόμαστε πολλές μεταμοσχεύσεις. Ωραία. Περνάμε στο θέμα του χρονοδιαγράμματος των περίοδων συνόδων. Κύριος Κέλλη. Καταρχήν να σας συγχαρώ γιατί χειριστήκατε πολύ σωστά αυτό το δύσκολο θέμα σήμερα. Εξηγήσατε την ερμηνεία του, του Προέδρου και επιμείνατε στις επιλογές του. Εγώ επειδή δεν είχα τη δική μου άποψη, ακολούσα τη δική σας. Δεύτερον, αυτό που ο κ. Σλάτο είναι πολύ σωστό. Χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε πιο γρήγορους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους να ερχόμαστε στο Στρασβουργό. Και χαίρομαι που το δεύτερο δρόμο της Φραγκφούρτης επίσης συμπεριληφθήκε. Νομίζω άλλωστε ότι θα βελτιωνόταν πολύ τα πράγματα στο Στρασβούργο αν οι ε, συνδέσει αυτή τη πόλη ήταν ίδιε τι εβδομάδε που εμεί συνερχόμαστε με αυτέ που δεν συνερχόμαστε. Θέλω να κάνω ε, μία εξήγηση, μία επεξήγηση για την έκθεση Μικολά, Μικολάσικα. Έχω στείλει και μήνυμα ότι θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για την μεταμόσχευση ανθρωπίνων οργάνων. Πολλοί πεθαίνουν κάθε μέρα γιατί έχουν πρόβλημα με κάποιο όργανο και γιατί δεν υπάρχει κανένα όργανο για να μεταμοσχευθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει του ασθενεί σε όλη την Ευρώπη με το θέμα των οργάνων και επομένω να σωθούν πολλέ ανθρώπινε ζωέ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα καλά συντονισμένο σύστημα δωρεά οργάνων και μεταμόσχευση. Θα ήθελα να τονίσω ακόμα μια φορά ένα πολύ σημαντικό σημείο που είναι και πολιτικής σημασίας, ειδικά την αρχή της εθελοντικής δωρεά τμήματων του ανθρωπίνου σώματος. Η έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και του Συμβουλίου της Ευρώπης λέει ότι σε πολλές χώρες του κόσμου δίδονται πάρα πολλά χρήματα από ανθρώπους ε, για δωρεές. μερικές φορές σκοτώνουμε ανθρώπους για τα όργανα τους, παραδείγματο χάρη στους Φαλούγκ στην Κίνα. Ορισμένες φορές ο ιατρικός κίνδυνος για τον δωρητή είναι πολύ ψηλός και η μεταμόσχευση γίνεται υπό κακές συνθήκες. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι το ψήφισμα που υιοθετήσαμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να συγχαρώ και τον εισηγητή του ψηφίσματος, τον κύριο Μικολάσικ. Τώρα, η κυρία Κοράτσα πρώτη. Σας ευχαριστώ. Εγώ είμαι κατά της απαγόρευσης της τρομβίνης. Γιατί γνωρίζουμε ότι ούτως ή άλλως η τρομβίνη δεν επιτρέπεται στα εστιατόρια και στις καντίνες και στους χώρους εστίασης. Πρέπει τώρα να φέρουμε τη συζήτηση στις σωστές διαστάσεις. Μιλάμε για τη θρομβίνη σε όλα τα είδη κρέατος. Ο ε, εκπρόσωπος Κομισιόν δήλωσε ότι η θρομβίνη δεν είναι επικίνδυνη για την υγεία και αυτό βασίζεται σε επιστημονικές αποδείξεις. Δεν πρέπει φυσικά να παραπλανούμε τον καταναλωτή. Απλώς πρέπει να επισημάνουμε ξεκάθαρα πάνω στα πακέτα κρέατος ότι το εν λόγω κρέας περιλαμβάνει περιέχει θρομβίνη. Ας μην ανοίξουμε, σας παρακαλώ, το κουτί της Πανδώρας. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Πρέπει να υπάρχει ελεύθερη επιλογή για τον καταναλωτή. Και δεν πρέπει να απαγορεύουμε ε, τρόφιμα, τα οποία δεν είναι επικίνδυνα. Απλώς χρειάζεται μια σωστή ε, επισήμανση. Όχι απαγορεύσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Δεν είναι κυρία Σόμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η διαδικασία σήμερα είναι καθαρά λαϊκιστική γιατί δεν προσανατολιζόμαστε σε επιστημονικά δεδομένα. Η θρομβίνη είναι φυσικό ένζυμο που περιέχεται στο αίμα, άρα και στο κρέας. Όλοι μας ε, έχουμε θρομβίνη στον οργανισμό μας. Το να απαγορεύουμε τη χρήση της σημαίνει ότι αυτό ανερούμεθα ως άχρηστο υλικό. Βεβαίως πρέπει να μην παραπλανούμε τους καταναλωτές Βεβαίως θα πρέπει να ενημερώνουμε για το τι ακριβώς είναι και γίνεται αυτό με το νέο κανονισμό για την επισήμανση των τροφίμων που θα, γίνει, θα συζητηθεί σε πρώτη ανάγνωση. Έχουμε πολλούς κανόνες κατά της παραπλανητικής διαφήμισης, την επισήμανση ειδικών προϊόντων και αυτό ελήφθη υπόψη και στα προϊόντα που χρησιμοποιείται η φθρομβίνη ως κόλλα. Υπάρχουν πολλά παρόμοια ένζημα που δεν απαγορεύονται και ε, χρησιμοποιούνται. Ευχαριστώ. Κυρία Βάις Κέρμπερ. Η προστασία των καταναλωτών με απασχολεί πολύ. Γι' αυτό τάσομαι κατά κάθε μορφής παραπλάνησης των καταναλωτών. Γι' αυτό αγωνίζομαι και στα πλαίσια του κανονισμού επισήμανσης τροφίμων για καλύτερη επισήμανση τροφίμων των ε, απομιμήσεων και καλό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την άποψη αυτή που στηρίζεται και από την Κομισιόν να τη δεχτεί. Σήμερα ψηφίσαμε για το συγκολλημένο κρέας, το οποίο σε τελευταία ανάλυση ε, πωλείται ως υψηλής ποιότητας προϊόν. Αυτό δεν επιτρέπεται, θεωρώ, ιδιαίτερα αν δεν το ξέρουν οι καταναλωτές. Ε, δεν ήταν εύκολο να αποφασίσω σήμερα. Η Κομισιόν πρότεινε μια καλύτερη επισήμανση, υποχρέωση επισήμανσης. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι παρόλα αυτά μπορεί να παραπλανηθεί ο καταναλωτής, διότι η θρομβίνη δύσκολα αποδεικνύεται και ανοιχνεύεται στο προϊόν. Χρησιμοποιείται, αλλά μετά μπορεί να μην δηλώνεται. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν επαρκεί υποχρέωση επισήμανσης εδώ. Γι' αυτό τάχθηκα υπέρ της απαγόρευσης των θρομβινών. Ευχαριστώ. Κυρία Μορβάη. E, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα προηγούμενα οκτώ χρόνια η... με τα κομμουνιστική Ουγγαρία ε, συνέχισε να αποδοπατεί τα δικαιώματα των πολιτών σχεδόν παντού διοργανώνονταν διαδηλώσεις, ταραχές που καταστέλλονταν με τη βία. Η υπηρεσία ε, προάσπισης του δικαίου προσπάθησε να παρέμβει και πολλά, πολλές δίκες έφτασαν στα δικαστήρια. Πολλές φορές έπρεπε να γίνει προσφυγή και στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί τώρα να χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για, για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου για να υποσκάψει ε, το ε, δίκαιο. Νομίζω ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εξεταστεί εντελεχώς. Θα πρέπει δηλαδή να διαμαρτυρηθούμε ε, κατά της έκθεσης ατόντο γιατί στην πραγματικότητα υπονομεύει τα δικαιώματα του ανθρώπου στην Ευρώπη έτσι όπως έχει το σύστημα τώρα. Είναι η ιστορική μας ευθύνη στην Ουγγρική Προεδρία να ανασχέσουμε και να ε, σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Μορβάη, εσεί ε, τοποθετήκατε επί τη έκθεση έτσι δεν είναι. Για την έκθεση Ατόντο νόμιζα ότι μιλούσαμε. Για την Ατόντο είχα ζητήσει το λόγο. Εσεί είστε πρόεδρε, Εσεί μου δώσατε το λόγο, τι να κάνω, εγώ ακολούθησα τι οδηγίε σα. Σωστό, σωστό. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Καταγράψαμε την ε, επεξήγησή σας εκεί που πρέπει. Συνεχίζουμε τη θρομβίνη. Κυρία Μορκουνέτε. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ λεπτό και ευαίσθητο αυτό το θέμα και προκάλεσε πολύ μεγάλη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, αλλά και στις κοινωνίες μας εν γέννη. Νομίζω ότι η απαγόρευση οποιοδήποτε προϊόντος, οποιοδήποτε προσθέτου, δεν είναι ένας σωστός τρόπος. Ε, ίσως ξεχνάμε το επιχείρημα ότι ο καταναλωτής πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέξει με βάση όλες τις πληροφορίες όμως, να του δίνουμε όλες τις σωστές πληροφορίες. Από την άλλη δηλαδή η διαχείριση της διαδικασίας δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Σε αυτή την εποχή όπου ο καταναλωτής έχει πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες και όπου υπάρχει μια μεγάλη έτσι, γνώση και αφύπνιση για αυτά τα θέματα, ε, οι διατυπώσεις γύρω από αυτά τα θέματα συχνά είναι απροσπέλευτες εντελώς. Πώς ένα άτομο επίσης μπορεί να ενημερωθεί σωστά όταν αγοράζει ένα προϊόν για να καταλάβει α, τι ακριβώς αγοράζει. Για να καταλάβει τα συστατικά. Αυτό είναι το βασικό. Νομίζω ότι υπάρχει λοιπόν όχι επαρκής διαβούλευση με το κοινό και όχι σωστά, α, σωστή πληροφορία. Δεν δίνεται σωστά η πληροφορία. ich denke, die europäischen Bürger Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δίκιο που λένε ότι ζητούν τίμια ε, τρόφιμα και τίμιους πολιτικούς. Σέβομαι τη γνώμη τους. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να γνωρούμε την κοινή γνώμη, ούτε να μιλάμε για λαϊκισμό. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρέπει να καταλάβουμε τα μηνύματα από τους πολίτες. Όταν οι εκλογείς μας, οι πολίτες θεωρούν ότι θέλουν γνήσια τρόφιμα και ότι το κρέας πρέπει να είναι γνήσιο και να μην είναι κολλημένο από υπόλοιπα, πρέπει να φροντίσουμε να μην ε, προσφέρεται τέτοιο κρέας. Ε, εγώ ψήφισα ε, υπέρ θεωρώντας τη θρομπίνη ένα τέτοιο μέσον. Κυρία Κάντενπαχ. Dank. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σήμερα ψήφισα ε, το ψήφισμα γιατί ο Επίτροπος δεν με έπεισε. Δεν θέλω με συγκολλημένο κρέας. Ακόμα και αν η θρομβίνη δεν βλάπτει την υγεία. Παρόλα αυτά ε, δημιουργεί ένα συμπιεσμένο κρέας το οποίο αυξάνει πολύ τον απικισμό από βακτήρια. Ε, έτσι λοιπόν χρειαζόταν μια σαφής, ένα σαφές μήνυμα προς τους καταναλωτές κατά της βιομηχανίας. Θέλουμε να τρώνε την μπριζόλα που θέλουν οι καταναλωτές μας και όχι κολλημένο κρέας. Η Κομισιόν δεν θα πρέπει λοιπόν να επιτρέψει την θρομβίνη. Ωραία. Περνάμε στην έκθεση Περελιό. Σχέδιο δράσης για τη μεταμόσχευση οργάνων. Περέγιο. Ποιος έχει το λόγο? Για την θρομβίνη θα ήθελα να μιλήσω, αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση για τα τρόφιμα ε, και προϊόντα κρέατος ε, δείχνουν μια στάση καταναλωτών. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει η επισήμανση να αποκλείει την παραπλάνηση των καταναλωτών. Αν χρησιμοποιείτε το ένζυμο θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον καταναλωτή. Αυτή είναι η βάση για λειτουργική και δίκαιη προστασία των καταναλωτών. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε ώστε ο πολίτης να έχει ε, τις κατάλληλες πληροφορίες για να λαμβάνει τις αποφάσεις του. Τώρα, ε, για το ζαμπόν το συγκολλημένο εδώ ε, θα πρέπει να ξέρει τι αγοράζει και αν θα το αγοράσει ο καταναλωτής. Ευχαριστώ πολύ. Λέω, περνάμε στο σχέδιο δράσης. Περνάμε στο σχέδιο δράσης για τη μεταμόσχευση οργάνων. Κυρία Οβίρ. Είναι ma ε, Καλωσορίζω αυτό το σχέδιο δράση, το υπερψήφισα, είναι ένα βήμα προ τη κατεύθυνση. Θα πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Χρειάζονται μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο, διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί και η δουλειά των κρατών μελών. Θα ενισχυθεί η ασφάλεια των οργάνων, των μεταμοσχεύσεων και, των, και η υγεία των ασθενών. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί γενικότερα το σύστημα και τα κράτη-μέλη θα έχουν πλέον την ε, δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτά τα 10 μέτρα προτεραιότητα στα εθνικά τους ε, σχέδια δράσης. Είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε αυτούς που δουλεύουν στον τομέα της ε, υγείας. Κυρία uh, Αυτά τα θέματα, αυτή η έκθεση με την έκθεση Μικολάσικ είναι παρόμοιες. Επομένως η εξήγηση που έδωσα για εκείνη την έκθεση ισχύει και εδώ. Ο κ. Μαστέλα. Πρόκειται για μία πρόοδο στην ε, πολιτική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προστασία των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων ε, είναι πολύ, βγαίνει ενισχυμένη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική σημασία του δικαιώματος που αναγνωρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σας παρακαλώ λίγο πιο αργά. Ναι, ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ θεωρούμε ότι είναι τεράστιας πολιτικής σημασίας το δικαίωμα που αναγνώρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το γεγονός ότι στέλνουμε στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης κάποιους αντιπροσώπους. Υπενθυμίζουμε ότι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και υπάρχει και στην ε, συστατική μας ε, συνθήκη. Επίσης θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της σύμβασης της νομολογίας του Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για να υπάρξει ένα νέο νομικό πλαίσιο με κατευθυντήριες αρχές στον τομέα των πολιτικών ελευθεριών, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων υπό το φως νέων ε, ολοκληρώσεων και λόγω της θέσης σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας καθώς και της υιοθέτησης του προγράμματος της Λισαβόνας. Επίσης, ε, υπάρχει και το πρόσθετο νομικό εργαλείο ε, και υπάρχει τη δυνατότητα να καταγγείλει κανείς στο Δικαστήριο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων το γεγονός ότι κάποιο θεσμικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιο κράτο μέλο αμελεί να πάρει κάποια συγκεκριμένη δράση υπέρ τη προστασία ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το άρθρο 1 τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Ε, εγγυόμαστε όχι μόνο την προστασία των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των αρνητών που διαμένουν στο εσωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όλου όσου ε, εντάσσονται στη δική μα δικαιοδοσία ακόμη και αν βρίσκονται εκτό τη επικράτειά μα. Ο κύριος Αντωνιώτσι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ είμαι υπέρ προσχώρηση προσχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, και η έκθεση Ατόντο είναι πολύ σωστή, αποτελεί ένα βήμα στην ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα βήμα ακόμη προς την πολιτική Ευρώπη. Ε, υπάρχει συνάφεια μεταξύ Ένωσης ε, και χωρών που ανήκουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης ε, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου. Αυτό θα αυξήσει την αξιοπιστία της Ένωσης απέναντι στις τρίτες χώρες και τέλος θα δείξει την στεναρή μας θέληση να εναρμονίσουμε σε νομοθετικό και νομολογικό πλαίσιο το θέμα των ελευθεριών και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νομική προσωπικότητα για πρώτη φορά και ελπίζω ότι η υπογραφή της ε, συνθήκης αυτής, της σύμβασης αυτής θα είναι ένα μόνο πρώτο βήμα για να συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το δέοντα τρόπο στις ε, μεγάλες διεθνείς διαπραγματεύσεις. Κυρία Μορβά, εσείς πήρατε ήδη το λόγο πριν. Ούτως ή άλλως την προηγούμενη παρέμβασή σας την καταγράφουμε και για αυτό το σημείο. Monsieur le Président, je suis un peu plus réservé que les collègues qui viennent de... Είμαι πιο επιφυλακτικό από τους προλαλήσαντες. Η ιδέα του ευρωπαϊκού δίκαιου να εμπίπτει στην δικαιοδοσία του, ε, Παγκόσμιου, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι ελκυστική. Θα έπρεπε το δικαστήριο να έχει δικαιοδοσία επί των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, δεν θα έπρεπε το ευρωπαϊκό δικαίωμα να ξεφεύγει από αυτή τη δικαιοδοσία. Πολύ δε περισσότερο που, για παράδειγμα, στην Γαλλία, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Συνταγματών μας, ε, το ε, διεθνές δίκαιο επικρατεί επί του εθνικού δικαίου. Όμως, υπάρχει ένα θέμα λεπικάλυψης πολλές ε, φορές το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν εφαρμόζεται άμεσα στις εθνικές νομοθεσίες αλλά απλώς μεταγράφεται μέσω ε, ενό δευτερογενούς δικαίου. Από την άλλη μεριά, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει δείξει σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και, και ιδιαίτερα αυτά που προκύπτουν από την των Θεμελιώδων Δικαιωμάτων. Συνεπώς, ενδεχομένως θα έχουμε αλληλεπικάλυψη διαδικασιών. Ιδιαίτερα αν ε, ιδρυθεί και συσταθεί και ένας μηχανισμός προδικαστικών ερωτημάτων. Ευχαριστώ. Περνάμε στη διάσκεψη για την αναθεώρηση του καταστατικού δρόμου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Δραματικά γεγονότα λαμβάνουν χώρα στην ε, Ταϊλάνδη. Συνεπώ, δικαιολογούμε να είμαστε ευαίσθητοι ω προ το ότι ε, θα πρέπει να μπορούν οι προτέτοι να ε, δικαστούν οπουδήποτε. Πλην όμω ακούσαμε πολλά πράγματα χτες στη συζήτηση και πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για το πρώτο διεθνέ ποινικό δικαστήριο μίλησαν για τις ε, Ναπάλμ στη Δρέσδη που έπεσαν χωρίς κανένα λόγο ε, για τη Χειροσύμα και τον Αγκασάκη ε, για αυτούς που δολοφόνησαν με μια σφαίρα πισόπλατα τους πολλούς αξιωματούχους και λοιπά και θα πρέπει και όλοι αυτοί να δικαστούν. Το απολογισμό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Ιουγκοσλαβία επίσης δεν είναι πολύ ικανοποιητικό. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Αποζημιώσεων, τα κράτη-μέλη θα πούν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αποζημιώσει όλους αυτούς που έχουν φύγει από τα σύνορα της κάθε χώρας. Είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μάλιστα άνθρωποι. Και πολλές ε, φορές πρέπει να πούμε ότι οι, οι τιμένοι μπορεί εξαιτία αυτού του καταστατικού να συνεχίσουν να μάχονται μέχρι τελευταία ε, αγώνα του αίματό του αντί να προβούν σε μια συμφωνία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το ψήφισμα για την διάσκεψη που θα αρχίσει τις εργασίες της αργότερα κατά τη διάρκεια του έτους περιλαμβάνει τις 138 χώρες που συνέστησαν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και το καταστατικό ε, που διέπει τις εργασίες του από το 2003 ήρθε η ώρα για αναθεώρηση, ιδιαίτερα τις μεταβατικές διατάξεις που ήταν αντικείμενο διαφωνίας το 2002. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, επικύρωσαν το καταστατικό. Όμως ε, οι εργασίες ε, του δικαστηρίου δεν λαμβάνει υπόψη κάποιους εταίρους όπως η παρουσία και Κίνα και σήμερα το Κοινοβούλιο καλεί τις χώρες αυτές να κυρώσουν το καταστατικό και να συνεργαστούν με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για γενοκτονία τον 21ο αιώνα που κατηγορούνται για ε, αδικήματα πολέμου δεν θα πρέπει να κρίνονται μόνο ηθικά αλλά να τιμωρούνται και από τον νόμο και κανείς δεν θα πρέπει να μείνει ατιμόρυτος. Τελειώσαμε τις επεξηγήσεις ψήφου. Διακόπτουμε μέχρι τις 3 το απόγευμα.